Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχω την τιμή να μπορώ να σας ανακοινώσω ότι το βραβείο Ζαχάροφ ε, το 2012 θα απονεμηθεί στους εξής. Ναστρίν Ζουτουντέ και Ζανάφα Πανάια από το Ιράν. Ε, οι δύο αυτοί, η Ναστρίν Σοτοντέ και ο Ζαφάρ Πανάη, λαμβάνουν το βραβείο με ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων και τους απονέμουμε το βραβείο αυτό εξ ονόματος όλων. Με αυτή την επιβράβευση εκφράζουμε το θαυμασμό μας για μια γυναίκα και έναν άντρα οι οποίοι δεν υπέκυψαν στον φόβο και την τρομοκρατία στο Ιράν και επιθυμούν η μοίρα της χώρας τους να είναι πάνω από την προσωπική τους μοίρα. Η Ναστρίνσο Του τέθηκε ε, στην προμετοπίδα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αντιφρονούντων. Λόγω λοιπόν αυτών των θαραλέων πράξεών της ε, η Νασρίν έχασε την οικογένειά της, απομακρύνθηκε από αυτήν ε, και δέχθηκε κατηγορίες όπως προπαγάνδα κατά του κράτους ή επίθεση κατά της εθνικής ασφάλειας. Καταδικάστηκε λοιπόν σε κάθριξη 12 ετών. Κυρίες και κύριοι, ο αγώνας για την ελευθερία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προσωπική αξιοπρέπεια, για την απαγόρευση των βασανιστήριων, για την ελευθερία έκφρασης σκέψης. Αν όλα αυτά αποτελούν επίθεση κατά της εθνικής ασφάλειας, τότε εμείς υποστηρίζουμε αυτούς που επιτίθενται κατά της εθνικής ασφάλειας μιας χώρας που δεν σέβεται κανένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το βραβείο προς την Νοστρίνσου Today είναι είναι μια κατάφορη, μια σαφής καταδίκη του καθεστώτος στο Ιράν. Ο Ζαφά Πανάη είναι ένας ε, από τους γνωστότερους ε, σκηνοθέτες. Ε, οι ταινίε του είναι η παρουσίαση μιας πλούσιας όμορφης χώρας και των κατοίκων της χώρας αυτής. Όπως σε όλα τα πορτρέτα που είναι και στα βιβλία του, ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζει τα καθημερινά προβλήματα, όχι μόνο τις αντιφάσεις και τις όμορφες πλευρές της χώρας, αλλά τα καθεστώτα είναι σαφές ότι δεν φοβούνται τίποτα περισσότερο από την πικρή αλήθεια που παρουσιάζεται ε, σε ταινίες και οπουδήποτε αλλού. Άρα δηλαδή ε, προσπάθησαν ε, και τους δύο να τους καταδικάσουν σε σιωπή αλλά και οι δύο είναι έκφραση των δικών μας των αξιών, των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε λοιπόν με δυνατή φωνή δεν είσαστε μόνοι σας και εύχομαι τον Δεκέμβρη να έρθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπους εδώ στο Στρασβούργο για να παραλάβουν τα βραβεία τους. Καλό λοιπόν τις αρχές του Ιράν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστεί δυνατή η μετάβασή τους στο Στρασβούργο. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους ε, που βρίσκονται εδώ ε, στο Στρασβούργο και συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία για τη βραβεία Ζαχάρου να δεχτούν τις ευχαριστήσεις μου. Εγώ από το 1994 είμαι εδώ στο κοινοβούλιο Κοινοβούλιο και έχω συμμετάσχει σε όλες τις ε, τελετές απονομής των βραβείων Ζαχάροφ με διάφορες ιδιότητες, αλλά ποτέ, μα ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε περίπτωση όπου η διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσει ομόφωνα. Ε, δεν υπήρχε καν αντιπρόταση. Πρώτη φορά λοιπόν απονέμεται ομόφωνα το βραβείο Ζαχάροφ. Τρία μόλις λεπτά χρειαστήκαμε σήμερα το πρωί για να λάβουμε την απόφασή μας και μου ήρθαν στο μυαλό άλλες συζητήσεις που είχαν προηγηθεί. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι σαφές ότι οι περισσότεροι εδώ στο Κοινοβούλιο επιθύμησαν να επιβραβεύσουν ε, την ε, κυρία και τον κύριο από το Ιράν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εσάς για την προσοχή σας. Ο κύριος Κέλλενεν ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κέλλενεν. Ευχαριστώ. Φυσικά και καλωσορίζω τη βράβευση αυτή με το βραβείο Ζαχάροφ και χαίρομαι ότι ήταν και ομόφωνη η απόφαση για την απονομή του βραβείου στους δύο εμ, γενναίους αυτούς αντιφρονώντες του Ιράν. Βέβαια, έχω βαθύτατες ανησυχίες για την κατάσταση στο Ιράν και ταυτόχρονα με την απονομή του βραβείου αύριο θα αποχωρήσει μια αποστολή ευρωβουλευτών για ε, κάποιες συζητήσεις με το καθεστώς του Ιράν. Πραγματικά είναι πονίδιστη αυτή η απόφαση να κάνουμε κουβεντούλες με τέτοια κυβέρνηση και τέτοιο καθεστώς. Βέβαια, δεν είναι διακομματική αυτή η αντιπροσωπεία. Απαρτίζεται κυρίως από αριστερούς ευρωβουλευτές και σίγουρα θα χειραγωγηθεί αυτή η επίσκεψη παρόλο που έχει στόχο να, να στηρίξει τους ακτιβίστες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ε, θα δώσουμε ανάμεικτα και συγκεχημένα μηνύματα δύο εβδομάδες μετά τις, ε, το λάθος που κάναμε να καταψηφίσουμε αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν. Ε, να στέλνουμε ευρωβουλευτές που θα πάνε να έχουν ψιλοκουβεντούλα και να πιούν και σαμπάνια με ηθήνοντες του Ιρανικού καθεστώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καλλινάν. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα δεν είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης. Γι' αυτό το ταξίδι, αυτή την επίσκεψη, αποφάσισε διάσκεψη των πρόεδρων και αποφάσισε επίσης ότι η αντιπροσωπεία θα ήταν καλό να το έχετε πει και αυτό προηγουμένως που λάβετε το λόγο. Αποφασίστηκε λοιπόν πριν από λίγα λεπτά τα αποφάσισε ότι θα λάβει χώρα αυτή η επίσκεψη θα λάβει μαζί της γραπτά τα συγχαρητήριά μας που θα επιδώσει, θα τα επιδώσει στους δύο αντιφρονούντες. Αν λοιπόν δεν το δεχτεί αυτό η ε, κυβέρνηση στο Ιράν, τότε στην περίπτωση αυτή δεν θα λάβει χώρα η επίσκεψη ή αν έχουν πάει εκεί επιτόπου θα αποχωρήσουν, θα φύγουν παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη να τοποθετηθείτε επί διαδικαστικού και όχι για το θέμα αυτό γιατί δεν προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη. Ό,τι ήταν απαραίτητο για το θέμα αυτό το είπα ήδη. Μικρόφωνο, παρακαλώ, ευχαριστούμε. Θα ήθελα να πω ότι στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλούνται ακτιβιστές να επισκεφτούν το Ιράν και να υποστηρίξουν επιτόπου τους ανθρώπους που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε αυτό που σας ανακοίνωσα. Βεβαίως ε, ε, θα μπορούσε κανείς ε, να προβληθεί λέγοντας κάτι διαφορετικό. Αυτό θελήσατε να κάνετε κύριε Κέλναν, δεν ξέρω αν ήταν σωστό. Εν πάση περιπτώσει το θέμα έχει κλείσει όπως ακριβώς αποφάσισε η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία. Ξεκινάω λοιπόν με την ψηφορία για έξι.